il Presidente. La seduta riprende ora. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση και με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να σας ανακοινώσω αυτό που μόλις έμαθα από τον τύπο και από ό,τι μάθαμε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει άρει την ε, ποινή της ε, κυρίας Σακίνε. Πρόκειται για μια απόφαση που ελήφθη λίγες ώρες πριν μετά από τον κοινό αγώνα που δώσαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό μας γεμίζει χαρά αλλά συνεχίζεται ο αγώνας μας για την αναθεώρηση της δίκης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα του παρελθόντος, δηλαδή να προασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο. Αρχίσουμε με τις εργασίες μας τα πρακτικά της ε, χθεσινής ημέρας και τα εγκεκριμένα κείμενα έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, τότε τα πρακτικά εγκρίνονται. Περνάμε τώρα στην προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο για τις εξαγωγές όπλων. Ο κύριος Κάρινς έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, έχετε λάβει ε, την προφορική ερώτηση και να σας εξηγήσω ελικοπτεροφόρα 200 μέτρων που μπορούν να μεταφέρουν 16 βαριά ελικόπτερα, 40 άρματα μάχης, εκατοντάδες οπλίτες. Ε, είναι ε, πολύ σημαντικά όπλα. Έχουν ε, επίσης και νοσοκομεία ε, εκστρατεία μέσα στα πλοία αυτά και αυτά τα τέσσερα σκάφη αποφάσισε η Γαλλία να τα πωλήσει στη Ρωσία χωρίς να ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από δύο χρόνια η Ρωσία επετέθηκε στη Γεωργία, γειτονική χώρα και δεν ε, τηρεί τα όσα επέτυχε η Γαλλία όταν μεσολάβησε. Ε, επίσης έχει όπλα κοντά στην Εστονία και κάνει ασκήσεις κατάληψης και εισβολής στις βαλτικές χώρες. Και ρωτώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είμαστε, τι τη χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έπληξε την Ελλάδα βαριά οικονομική κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε την επιλογή να βοηθήσει την Ελλάδα ή να την αφήσει να καταβυθιστεί. Ε, έδειξαν αλληλεγγύη βοηθώντας την Ελλάδα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, γιατί ήξεραν ότι αν επιδεινωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα θα επιδεινωθεί και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τομέας λοιπόν της εξωτερικής ασφάλειας δεν είναι εξαίρεση. Και εδώ και στη συνθήκη έχουμε ε, δεσμευτεί να δρούμε με τρόπο αλληλέγγυο. Πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανησυχούν. Για ποιο λόγο τώρα θέλει η Ρωσία να χρησιμοποιεί τέτοια πολεμικά πλοία. Ωραίε, καλέ και σημαντικέ είναι οι γαλλικέ θέσει απασχόληση, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να γίνει τη βάρο τη εθνική ασφάλεια άλλων κρατών μελών. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να απορρίψετε την πώληση όπλων σε τρίτες χώρες αν δεν συζητηθεί στο Συμβούλιο αυτό το θέμα και αν δεν έχουμε εγγυήσει ότι αυτά τα πράγματα θα βοηθήσουν, θα βελτιώσουν την κατάσταση ασφαλείας και δεν θα την επιβαρύνουν. Ευχαριστώ κύριε Κάριντς. Δίνουμε τώρα το λόγο στον αναπληρωτή Υπουργό εξ ονόματος του Συμβουλίου, τον κύριο Τσάστεν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι ε, Ευρωβουλευτές, ε, Είμαι ευτυχής για την ευκαιρία που μας δίνεται απόψε για να εξετάσουμε τις εξαγωγές οπλισμών. Επειδή είπατε εκπρόσωπος η κυρία Άστον δεν είναι δυνατόν να είναι παρούσα σε αυτή τη συνεδρία, συζήτησα από την Προεδρία να την αντικαταστήσει για αυτή τη συζήτηση και γι' αυτό θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μια σειρά από ερωτήσεις που λάβαμε για το θέμα αυτό. Όπως γνωρίζετε εδώ και πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των εξαγωγών όπλων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ο στόχος είναι σαφής, Θέλουμε να εμποδίσουμε τις εξαγωγές στρατιωτικής τεχνολογίας που μπορούν να χρησιμοποιηθεί για όχι καλούς σκοπούς όπως την καταστολή στο εσωτερικό μιας χώρας ή σε διεθνές επίπεδο. Πριν από 10 χρόνια το Συμβούλιο υιοθέτησε έναν διοντολογικό κώδικα σε θέματα εξαγωγής όπλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδεται μια σειρά από κριτήρια για την εξαγωγή σημαντικών όπλων. Αυτός ο κώδικας αντικαταστάθηκε το 2008 από μια κοινή θέση η οποία καθιέρωσε μια σειρά από νέα στοιχεία Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον έχει σήμερα, το, έχει, διαθέτει το, το πιο πλήρες καθεστώς ελέγχου πλεισμών στον κόσμο. Η, νομικά, ο νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα τη κοινή θέση εγγυάται ότι τα κράτη-μέλη θα προβαίνουν σε εξαγωγέ όπλων με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο. Η κοινή θέση έχει σαν σκοπό να συντονίσει αποτελεσματικά τις εθνικές πολιτικές σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της εξαγωγής όπλων μέσω μηχανισμών ενημέρωσης και διαβούλευσης για τι αρνήσει. και σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό όταν ένα κράτο μέλο σκέφτεται να δώσει άδεια εξαγωγή για μία συναλλαγή που ε, εξισούται με μία συναλλαγή που την αρνήθηκε προηγουμένω άλλο κράτο μέλο, πρέπει να διαβουλευτεί με αυτό το τελευταίο κράτο μέλο και να ενημερώσει όλα τα υπόλοιπα για την οριστική του τελική απόφαση. Το κράτο μέλο που χορηγεί άδεια για μία συναλλαγή που την αρνήθηκε άλλο κράτο μέλο, πρέπει να δικαιολογήσει την απόφασή του ενώπιον όλων των κρατών μελών. Για να απαντήσω λοιπόν στα ερωτήσεις σχετικά με τις διαβουλεύσεις, η κατάσταση είναι σαφής. Η κοινή θέση προβλέπει μια διαβούλευση, συστηματική διαβούλευση, μόνο στις περιπτώσεις όπου μια ταυτόσιμη συναλλαγή ε, ε, δεν έγινε δεκτή, ε, δεν, δεν της χορηγήθηκε άδεια. Κατά κανόνα τα γενικά τα κράτη-μέλη στα πλαίσια των δομών του Συμβουλίου ανταλλάσσουν τακτικά απόψεις και πληροφορίες για τον έλεγχο των οπλισμών και ειδικότερα για τα, τους ε, ονομαζόμενους ευαίσθητους προορισμούς. Ζητούν τα κράτη-μέλη τη Συμβουλή άλλων μελών του Συμβουλίου για οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία δημιουργεί ανησυχίε και για την οποία θα υπάρχουν αμφιβολίες. Αυτές οι ανταλλαγές πληροφοριών που είναι τακτικές αποτελούν σημαντικό στοιχείο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τον έλεγχο των οπλισμών. Το 2009 η διαβουλεύση μεταξύ κρατών μελών σας πληροφορώ, κάλυψαν 14 τρίτε χώρες προορισμού. Τα κράτη-μέλη του έδωσαν στοιχεία που τους τα είχαν κάνει να αποφασίσουν είτε να χορηγήσουν ή να αρνηθούν άδεια, την άδεια εξαγωγής προς αυτούς τους προορισμούς. Κύριε Πρόεδρε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, τον έλεγχο και την διαδραστική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών για να είμαστε βέβαιοι, πρωτού αποφασίσουμε να εγκρίνουμε ή να ε, απορρίψουμε την εξαγωγή όπλων. Σε μια άλλη απάντηση θα καλύψω οποιοδήποτε σημείο θα θέλατε να θίξετε στη διάρκεια της απογευματινής αυτής Grazie, συζήτησης. Ευχαριστούμε κύριε Σαστέλ. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπρόκ για δύο λεπτά. Που νομίζω ότι είναι απόν. Συνεπώς δίνω το λόγο στον κύριο Γκουαλτιέρη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μιλάμε για ενίσχυση της ε, βιομηχανίας και της ευρωπαϊκής άμυνας και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα κοινό αμυντικό σύστημα. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στον τομέα της άμυνας και να ακολουθήσουμε και τις διεθνείς μας δεσμεύσεις. Γι' αυτό υπάρχει και η κοινή θέση του Δεκεμβρίου του 2008, η κοινή θέση έτσι ώστε να δούμε ποια είναι η στάση μας έναντι των τρίτων χωρών. Μεταξύ αυτών των διαδικασιών δεν υπάρχει ένας γενικευμένος μηχανισμός διαβουλεύσεων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε στην ενίσχυση της συνεργασίας στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Θεωρούμε ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος και είναι δυνατόν να εισαχθούν ακόμα πιο δεσμευτικοί μηχανισμοί, αλλά θα έπρεπε η σύγκληση που προβλέπεται από το άρθρο 7 να μην παραμείνει κενό γράμμα και να δούμε ποια είναι η θέση μας ως προς τις εξαγωγές οπλισμών. Το ΕΛΚ θεώρησε ότι δεν θα πρέπει να παραμείνουμε στις γενικές γραμμές του σχεδίου, αλλά ας λέγαμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θεωρούμε ότι η πώληση όπλων από τη Γαλλία στη Ρωσία δεν αντιτάσσεται στην πολιτική μας, ίσα ίσα οδηγεί σε περαιτέρω δεσμεύσει στις διμερείς σχέσεις Γαλλίας-Ρωσίας και θα πρέπει να συζητηθεί, το, να το όλο θέμα και να τεθεί σε ευρωπαϊκή διάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί αρκεστήκατε στο χρόνο σας και κερδίσετε και πέντε δευτερόλεπτα. Βλέπω ότι στο μεταξύ έφτασε ο κύριος Μπροκ με μικρή καθυστέρηση και οπωσδήποτε θέλουμε να τον ακούσουμε, άρα με μεγάλη χαρά του δίνω τον λόγο. Ζητώ συγγνώμη, είχα ομάδα επισκεπτών, αλλά αμφιβάλλω ε, δεν μπορεί να ζήσει ε, το παρόν ακροατήριο αν δεν με ακούσει και εμένα. Μια παρατήρηση. Αυτή είναι παλιά ιστορία. Ποια είναι η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, για ποια θέματα και στη διακυβερνητική και στη συντακτική συνέλευση δεν καταφέραμε να βάλουμε στην κοινή ευρωπαϊκή αρμοδιότητα το εμπόριο όπλων. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε έτσι ώστε ο κώδικα συμπεριφορά και ρυθμίσει του Συμβουλίου του 2008 κάπω να γίνει δεσμευτικός και να συνδέεται με την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Θέλω να πω ότι για μένα είναι σαφές ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο δεν ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να έχουμε τόσο λίγες επαφές μεταξύ διαφόρων κρατών μελών, έτσι ώστε ορισμένα κράτη-μέλη να έχουν την αίσθηση ότι οι εξαγωγές όπλων σε τρίτους έρχονται εις βάρος τους και ε, διακυβεύουν τη δική τους εθνική ασφάλεια. Δεν ε, λέω ε, ότι έχουν δίκιο ή άδικο. Αν θέλετε αυτό δεν είναι και κάτι που μας ενδιαφέρει, είναι περίπου αδιάφορο. Θα πρέπει ε, να βρεθεί ευρωπαϊκή λύση. Και τρίτον, πιστεύω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία και για αυτά τα θέματα. Ας πούμε και μέσω του αμυντικού οργανισμού για να ε, δούμε και για λόγους βιομηχανικής πολιτικής τι πρέπει να κάνουμε. Και στις εξαγωγές αλλά και στην έρευνα, στο σχεδιασμό, στην παραγωγή ε, των εξοπλισμών να συνεργαζόμαστε περισσότερο και προμήθειες τις αμυντικές. Γιατί η αμυντική βιομηχανία έχει μεγάλη σχέση με ανεξαρτησία. Αν δεν έχουμε τίποτα και τα αγοράζουμε όλα από τρίτε χώρε, έχουμε και πολιτική εξάρτηση και εξάρτηση ασφαλεία. Αυτό έχει να κάνει και με την ελευθερία μα. Δεν είναι μόνο οικονομική σκοπή. Χωρί αυτή να είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Όλα αυτά θα τα πρέπει να βλέπουμε σε ένα συνολικό πλαίσιο. Γι' αυτό θα πρέπει να κοινωνικοποιηθεί περισσότερο και να μην έχουμε τέτοιες παρεξηγήσεις και να αισθάνονται ότι αδικούνται ή ότι απειλούνται ορισμένε χώρε μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μπροκ. Ουδής αναντικατάστατος, αλλά σίγουρα εσείς συνεισφέρετε κατά πολύ σε αυτή τη συζήτηση. Ο κύριος Βαν Μπάλεν έχει το λόγο για δυόμιση λεπτά. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σαφής. Και ε, εσείς μπορείτε και οι Γάλλοι μπορούν να υπερασπίζονται τον εαυτό τους. Ε, δεν θα πρέπει να εξάγουμε όπλα διάκριτα, αυτό λέει η ομάδα των φιλελευθέρων, δεν θα πρέπει να εξάγουμε όπλα σε περιοχές όπου έχουμε στίες πολέμου ή εντάσεων. Να περιοριζόμαστε. Και αν δεν έχουμε δεσμευτική ρύθμιση για τις εξαγωγές όπλων. Αυτό σημαίνει ότι τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ε, ίσους κανόνες παιχνιδιού και ανταγωνίζονται και διαγωνίζονται μεταξύ τους για προμήθειες και για παραγγελίες. Οπότε, ο μόνος τρόπος να λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι να έχουμε κάποια δεσμευτική ρύθμιση, κοινή ρύθμιση στην Ευρώπη και συμφωνώ με τον κύριο Μπροκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντικό το θέμα και ευχαριστώ τους συναδέλφους που αντιλαμβάνονται τις προβληματισμούς, τις ανησυχίες της περιοχής μου σε ό,τι αφορά αυτή την ε, απόφαση για τα Μιστράλ της Γαλλίας. Μιλάμε για ένα δεσμευτικό κείμενο εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν επαρκεί όπως τόνισε και ο συνάδελφος των φιλελευθέρων. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μεγάλη ευθύνη. Είμαστε υπεύθυνοι για το 1 τρίτο του εμπορίου όπλων. Εάν θεωρούμε ότι είναι στρατηγικό εταίρος η Ρωσία και μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τη χώρα αυτή για, για στρατιωτικά θέματα. Το ερώτημά μου είναι γιατί χρειάζονται ένα οπλικό σύστημα επιθετικό για να εξασφαλίσουν κάποιο σύστημα καλής διαχείρισης και διακυβέρνησης στο Αφγανιστάν. Ασφαλώς όχι θέλουν να προστατεύσουν τα δικαιώματα των, των, των μειονοτήτων στο Κυργιστάν. Προφανώς όχι και δεν τους χρησιμεύει το Μιστράλ ε, σε μια τέτοια περίπτωση διότι δεν είναι δυνατόν να φτάσει σε αυτές ε, τις περιοχές μπορεί ε, να επηρεάσει 8 κράτη-μέλη γύρω από τη Βαλτική και την κατάσταση ασφάλειας της Πολωνίας, της Γερμανίας, καταλήγοντας τη Λιθουανία, την Λετωνία και την Εστονία. Συμφωνώ με τον κύριο Γκουετιέρη ότι η συνεργασία με τους στρατηγικούς εταίρους μας είναι κάτι το καλό, το χρήσιμο. Αλλά υπάρχουν και άλλους τομείς συνεργασίας με τη Ρωσία από ότι ο τομέας των ε, οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Υπάρχουν ε, τα αυτοκίνητα, τα οχήματα, συνεργασία μεταξύ πυροσβεστικών υπηρεσιών. Οι Ρώσοι πυροσβέστες είχαν προβλήματα το καλοκαίρι ε, όταν άρχισε, εξέσπασε μια πυρκαγιά σε μια έκταση του μεγέθους του Βελγίου. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να τα ξανασκεφτούμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Παρακαλούσα τους ομιλητές να μην υπερβαίνουν το χρόνο που τους έχει απονεμηθεί. Βαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Εμείς προσδίδουμε μεγάλη σημασία στην εθνική κυριαρχία και εμείς θα αποφασίσουμε κατά πόσο θα προβούμε στην αδειοδότηση εξαγωγής όπλων. Δεν πρόκειται για μια κοινή ευρωπαϊκή θέση, δεν είναι ένα θέμα που αφορά αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως τα κράτη-μέλη που είναι καθαροί εξαγωγή θα πρέπει να λάβουν υπόψη μεταξύ άλλων και την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Θα πρέπει να γνωρίσουμε την ευαίσθητη κατάσταση που ισχύει και στη Μαύρη Θάλασσα και στις Βαλτικές χώρες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη γεωργία και τα παράκτια της ε, ε, Μαύρης Θάλασσας, διότι η Τουρκία και η Βουλγαρία είναι κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν και ε, αμφίβια πολεμικά οπλοστάσια τα οποία θα μπορούσαν να εξαχθούν. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την ε, σύμβαση που ισχύει για τα οπλικά συστήματα που μπορεί να συνέλθει κάθε έξι εβδομάδες στις Βρυξέλλες. Είναι το σωστό φόρμ για να συζητηθεί ε, το θέμα και όχι στο Στρασβούρο στην Ολομέλεια. Ευχαριστούμε τον κύριο Βανόρντεν. Λέζινγκ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Το έτος 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη στρατηγική της Λισαβόνας είχε λέει ως στόχο μέχρι το 2010 να είναι η πρώτη οικονομική δύναμη του κόσμου. Αυτό δεν το πετύχαμε σε πολλούς άλλους τομείς, αλλά εξαίρεση αποτελεί η εξαγωγή όπλων. Από το 2005 μέχρι το 2009 τα κράτη-μέλη ξεπέρασαν και τις Ηνωμένε Πολιτείες και είναι παριθμόν ένα εξαγωγέας όπλων στον κόσμο. Εγώ θεωρώ άκρος ε, προβληματική αυτή την κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς ε, νομικά δεν είχαμε δεσμευτικό κώδικα συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων και προέβλεπε περιορισμό υποτίθεται ε, στις εξαγωγές με όρους και προϋποθέσεις αλλά αυτό ήταν σκέτη φούσκα. Το Δεκέμβριο του 2008 ε, αυτός ο κώδικας έγινε κοινή θέση του Συμβουλίου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε ακόμα αποτελεσματικές σκυρώσεις. Παράδειγμα, η Γερμανία ήδη πολύ πριν το 2008 το έχει εγκρίνει αυτός δεσμευτικά, αλλά στο μεταξύ είναι παριθμόν τρία εξαγωγές όπλων στον κόσμο και εξάγει στην ε, Σαουδική Αραβία ή στο Πακιστάν όπλα που είναι περιοχές σε κρίση. Επιπλέον οι εκθέσεις των κρατών μελών προς το Συμβούλιο της Ένωσης δεν είναι ενιαίες και πολύ συχνά δεν είναι και διαφανείς. Επιγόντως χρειάζεται εδώ εναρμόνιση έτσι ώστε όλοι να μπορούν να αποδεικνύουν τι όπλα εξάγουν, σε ποιον και να ε, λογοδοτούν και ε, με κριτική σκέψη. Δυστυχώς προς την κατεύθυνση αυτή ε, της ομοιογένειας και της εναρμόνισης δεν υπάρχει. Αφήστε δε που εγώ αμφισβητώ και το ηθικό σκέλος της υπόθεσης αυτής. Πάντως είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει πόρο από τις ε, σωστές κινήσεις που θα έπρεπε να κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λέζιν, δυνάμει της ε, διαδικασίας της μπλε κάρτας, ο κύριος Βανόρτεν θα ήθελε να σας υποβάλει μία ερώτηση. Εσείς δέχεστε την ερώτηση από τον κύριο Βανόρτεν. Έχετε το λόγο κύριε Βανόρτεν. Uh, Κυρία Λόσινγκ έπεσε σε μια παγίδα που συχνά ακούγεται σε αυτό το κοινοβούλιο και αλλού. Αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή, εξαγωγές όπλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξάγει όπλα, δεν έχει αμυντική βιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενόπλες δυνάμει. Όλα αυτά ανήκουν στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ορολογία η οποία, ε, όπως οι ε, εξαγωγέ όπλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι που δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. λέει παρόλα. Χωρίς μικρόφωνο. Δεν ακούσαμε τι είπατε. Χωρίς μικρόφωνο μίλησε κύριε Είπα ότι τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είπα Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε με τη συζήτηση και δίνουμε το λόγο, το λόγο στον κύριο Κάμπελ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ε, εξαγωγής όπλων είναι αποτέλεσμα της ευρύτερης στατικοποίησης την συνθήκη της Αβώνας. Ο Τόνι Μπλερ πριν από λίγες μέρες είπε δημοσιογράφος ήθελε να δει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύσσει, ε, να, αποκτήσει, να αποκτήσει στατιωτικό χαρακτήρα μέσα σε από πού θα παίρνει τα όπλα της Ευρωπαϊκή Ένωση και πού θα τα πουλάει. Ο εξοπλισμός για, που κατασκευάζεται για τον ε, στρατό τον Ευρωπαϊκό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι σύμβατος με εκείνο των Ηνωμένων ε, Πολιτειών. Επίσης θα, κλειστεί, θα κλειστούν οι εξαγωγές προς την Αμερικανική αγορά και από την Αμερικανική αγορά προς την Αγγλική αγορά με, με αποτέλεσμα να χαθούν πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης και αυτό θα είναι ε, μια τεράστια οικονομική ζημία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ώρα, Για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ πρόεδρε αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο δίλημα όλες οι βιομηχανίες. Το κόστος είναι ιδιαίτερα ψηλό και συνεπώς δεν μπορούν όλες οι χώρες να παράγουν όπλα για ίδια χρήση. Άρα θα ήταν δελεαστικό να προβάλλουν ορισμένες χώρες μία πολιτική εξαγωγής όπλων και αυτό είναι, θα οδηγούσε από μία δεοντολογικά καλή πολιτική σε μία δεοντολογικά κακή. Ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει θέμα αντιμετώπισης εξωτερικού εχθρού. Οι χώρες που δεν έχουν σωστή τήρηση ανθρωπιστικών δικαιωμάτων, όπως το Ιράν, και άλλες χώρες, ιδιαίτερα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πρέπει να διαθέτουν αυτά τα όπλα. Αλλά όταν πρόκειται για υπεράσπιση έναν διεξωτερικού εχθρού, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να φέρουν αυτά τα όπλα. Επίσης, ε, θα πρέπει να πολλούνται μικρά όπλα και όχι όπλα μαζικής ε, καταστροφής. Η ΕΠΑ ΕΕ σταθεροποίησαν τον κόσμο και οδήγησαν σε μάλλον ανέλαβαν παράνομους πολέμους με όπλα και μαζική καταστροφή στο Ιράν δεν έχει επιτεθεί στις γείτονες ε, χώρες. Δηλαδή δεν επιτέθηκε στον, ε, παρά στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Όμως δεν θα έπρεπε να φέρουν ε, όπλα πάντα, αλλά θα μπορούσαν να έχουν μία πυρηνική ασπίδα για να μην τύχουν επίθεσης από τρίτους. Ο κύριος Τάνοκ θα ήθελε να υποβάλει μία ερώτηση προς τον κύριο Μπρόνς. Εάν ο κύριος ε, Μπρόνς μπορεί και θέλει να αποδεχτεί βέβαια αυτή την ερώτηση. Κύριε Τάνοκα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, δεν παρεμβαίνω σε συζητήσεις με άλλον ε, Βρετανό Ευρωβουλευτή αλλά κατηγορήθηκε κράτος μέλος να φυλακίζει ανθρώπους επειδή είχαν διαφορετική άποψη. Μπορεί να επικρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν νομίζω ότι υπάρχει ευρωπαϊκό κράτος μέλος που να φυλακίζει κάποιον για τις πολιτικές του πεπιθήσεις. Γιατί οι άνθρωποι θα... Γιατί αλλιώς... Πώς αλλιώς θα βρισκόταν ορισμένοι άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα Ποια χώρα, ποια χώρα φυλακίζει ανθρώπους για τους, λόγω πολιτικών πεπιθήσεων. Κάποιος παρεμβαίνει χωρίς μικρόφωνο από την αίθουσα. Θέλετε να απαντήσετε κύριε Μπρόνς. Θέλετε να απαντήσετε κύριε Μπρόνς. Κύριε Μπρόντς. Ουγγαρία στο προηγούμενο καθεστώς φυλάκισε αρκετά άνθρωπα για πολιτικούς λόγους. Υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που φυλακίζουν ανθρώπους ε, διότι, δεν συμφωνούν με τις απόψεις τους. Αλλά δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να ε, φυλακίζονται άτομα κυρίως όταν οι εκφράζουν πεπιθήσεις κατά της εξαγωγής και κατά το εμπόριο όπλων. Δίνουμε τώρα το λόγο στους άλλους ομιλητές. Αρχίζοντας από τον κύριο ε, Γκάλερ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να κάνω μεγάλη τιμή στον προλήσαντα και να αναφερθώ στην ομιλία του, αλλά είπε κάτι σωστό στην αρχή. Ότι για πολλά κράτη-μέλη που έχουν ε, μικρή πολεμική βιομηχανία αμυντική βιομηχανία είναι πολύ ακριβό να παράγουν τα δικά τους όπλα ο καθένας. Εγώ καταλήγω σε άλλο συμπέρασμα από τον ίδιο ότι με τον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Οργανισμό και με κοινά προγράμματα ε, προμηθειών αμυντικών ε, και οπλικών συστημάτων ε, θα μας βγαίνει πιο φτηνά. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για την τοποθέτησή του και θεωρώ πολιτικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχουμε την ευκαιρία να πούμε σήμερα ότι παγκοσμίω έχουμε τα πιο σύγχρονα και πιο νομικά δεσμευτικά δεσμευτικά κριτήρια για τις εξαγωγικέ όπλων. Κανείς δεν μπορεί να προσάψει τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί να είναι περήφανη γι' αυτό. Και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για στο Συμβούλιο σχετικά με αυτό. Μας εξηγήσατε σε ποιες περιπτώσεις η διαβούλευση ε, γίνεται. Και αυτό γίνεται όταν ε, απορρίπτονται κάποιες συμβάσεις σε μια χώρα, ενώ σε κάποια άλλη εγκρίνονται. Πού γίνονται αυτές οι συζητήσεις, σε επίπεδο ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και μόνο. Ή μήπω έχει συζητηθεί ποτέ αυτό και σε επίπεδο πολιτικό, ενώ υπουργών στο Συμβούλιο. Θα με ενδιέφερε. Έχω να πω πολλά ακόμα, δυστυχώς χρόνο δεν έχω. Τώρα δίνουμε το λόγο στον κύριο Παλέτσκης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, είπαν ότι ε, απαντώντας ότι η ερώτηση του ΕΛΚ περιέχει και κάποια ενίγματα και δεν διατυπώνεται, χωρίς να διατυπώνεται σαφώς το πρόβλημα. Μεγαλύτερη συμφήνεια θα ήταν χρήσιμη. Πρέπει να παραδεχθούμε ωστόσο ότι κάποιες χώρες Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες για τα στρατιωτικά θέματα διότι αισθάνονται πιο ανασφαλή από τα παλαιότερα ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 8 Δεκεμβρίου 2008 η το κοινό ψήφισμα του Συμβουλίου καθιερώνει κάποιους κανόνες σε θέματα εξαγωγής όπλων. Οι μεγνωγνώμονες δέχονται ότι η χώρα που αναφέρθηκε σήμερα, η Γαλλία δηλαδή, δεν ξεπέρασε τα όρια τα οποία είχαν προβλεφθεί. Αυτό σημαίνει ωστόσο ότι δεν θα έπρεπε να ε, ε, επεκτείνουμε, να παρατείνουμε τα όρια αυτά εφόσον προωθούμε μια κοινή θέση για αυτά τα θέματα. Πρέπει να συνεργαζόμαστε όλο περισσότερο στα θέματα των οπλισμών όπως και σε άλλους τομείς με άλλα κράτη-μέλη αλλά πρέπει να και άλλες χώρες, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επικρατεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από ό,τι συμβαίνει σήμερα διότι με τον τρόπο αυτό, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή δυσπιστία ανάμεσα στα παλιά και τα καινούρια κράτη-μέλη. Κάτι που πρέπει να αποφύγουμε. Πρέπει να επικοινωνούμε μεταξύ μας πιο συχνά για να αποφύγουμε να ε, ε, κατηγορούμε ημέν τους δε. πρέπει να, αποφύγουμε την επίδειξη δυνάμεων που είχε επικρατήσει πριν από μερικές δεκάδες χρόνια στην, Ευρώπη να συζητούμε αντίθετα με επικοδομητικό τρόπο διότι μόνο έτσι θα καταλήξουμε σε κάποιο χρήσιμο αποτέλεσμα. Ο κύριος Σαρνέτσκι έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ωραία λόγια ακούμε εδώ για την εμπιστοσύνη, για τη συνεργασία, αλλά νομίζω ε, στην πραγματικότητα και στην ουσία όταν πρόκειται για τις εξαγωγές όπλων βρισκόμαστε μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα. μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα πρότυπα, τις προδιαγραφές, την ηθική, τη διοντολογία που αναφέρουν πολλοί εδώ. Τις τελευταίες μέρες ξαναείδαμε αυτό το φαινόμενο. Η Γαλλία πουλάει σκάφη Μιστράλ στη Ρωσία. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ε, πώληση αυτή, γιατί η Ρωσία έχει ξεκινήσει μια διαδικασία πάρα πολύ ειδική και συγκεκριμένη ε, διαγωνισμών αλλά θα ολοκληρωθεί αυτή η πώληση και μόλις δήλωσε ένας Ρώσος ναύαρχος ότι αν η Ρωσία ε, διέθετε αυτά τα πλοία κατά τη διάρκεια της επίθεσης της στη Γεωργία, ο πόλεμος κατά της Γεωργίας δεν θα διαρκούσε τέσσερις ημέρες, αλλά τέσσερις ώρες. Ωραία. Ε, τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να πουλάνε τέτοια όπλα σε τέτοιες χώρες που θα τα χρησιμοποιήσουν ε, για ε, σκοπό επιθετικό και όχι αμυντικό. Η Γεωργία δεν μπορεί να προμηθευτεί ε, αμυντικά όπλα, διότι τις το αρνούνται. Διπλές προδιαγραφές. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Χουντής, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαβάζοντας την κοινή θέση και τα κριτήρια τα οποία πρέπει να τηρούνται από τις χώρες στις οποίες εξάγονται, χρήματα, εξάγονται όπλα, συγγνώμη, μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα του ισραήλ ένα κράτο που δεν σέβεται το διεθνέ δίκαιο που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει εισβάλει στη γάζα και εδώ αγαπητοί συνάδελφοι και σε αυτού που υπέβαλαν την ερώτηση δεν είδα από την πλευρά του με βάση τα τελευταία γεγονότα να υψωθεί μια φωνή ανάμεσα στι άλλε κυρώσει που πρέπει να επιβληθούν στο ισραήλ που δεν σέβεται αυτά τα κριτήρια που κατά τα άλλα έχουν τεθεί με την κοινή θέση να υπάρχει και η κύρωση μη εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού μη εξαγωγή όπλων ο αρχικό ομιλητή αναφέρθηκε με την έννοια τη πολιτική αλληλεγγύη τη Ευρώπη, στο παράδειγμα τη Ελλάδα. θέλω να σα θυμίσω κύριοι συνάδελφοι ενώ στην κοινή θέση στο κριτήριο 8 όταν θέλει να εξάγει μια χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια άλλη παίρνει υπόψη και την οικονομική δυνατότητα τη χώρα που πρέπει ή θέλουμε να εξάγουμε όπλα στην περίπτωση της ελλάδας η θελουμε να εξαγουμε οπλα στην περιπτωση τη ελλαδα η γαλλια και η γερμανία ενώ βρίσκεται σε άσχημη οικονομική κατάσταση ενώ υφίσταται πολλαπλού ελέγχου, ενώ περικόπτονται συντάξει ε, μισθοί κτλ πιέζουν για να εξασφαλίσει την πολιτική του υποστήριξη επαναλαμβάνω η γερμανία και η γαλλία να αγοράσει όπλα από αυτού. η θέση λοιπόν αυτή είναι υποκριτική και δείχνει ότι μέσα σε όλη αυτή τη λογική το πρόβλημα είναι ότι κυριαρχούν τα κέρδη των στρατιωτικών βιομηχανιών και όχι μια θέση αρχή που πρέπει να ακολουθεί η ευρωπαϊκή ένωση φιλιρινική και όχι επίλυση των διαφορών με στρατιωτικού τρόπου. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Πασκά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης που βρουν σε αυτό το τομέα. Παράγουν, κατασκευάζουν ε, όπλα. Και βεβαίως οι χώρες αυτές είναι ε, πρόσδεκτες στον υπόλοιπο κόσμο. Το εμπόριο όμως είναι εντελώς διαφορετικό σε αυτό το τομέα σε σχέση με άλλα αγαθά ως προς την ε, κοινή θέση άμυνας και ασφάλειας, διότι αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει με βάση ειδική εθνική αδειοδότηση για την εξαγωγή στρατιωτικού υλικού δηλαδή ή για να μεταφερθεί ενδοκινοτικά. Για όλα αυτά χρειάζεται ειδική άδεια, η οποία διέπεται από λεπτομερείς κανόνες και επίσης σοβαρή εποπτεία, αυστηρή εποπτεία. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή πρόκειται για ένα εξειδικευμένο θέμα, θα πρέπει να υπάρξει μια εξατομικευμένη προσέγγιση του θέματος απλώς να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις στην άμυνα και την ασφάλεια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντανζό έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα αναφερθώ σε τρία σύντομα σημεία για αυτό το θέμα. Πρώτον, επειδή αναφέρθηκε η θέση της Γαλλίας ε, ό,τι αφορά την πωλή στον Μιστράλ και θα, θα σας θυμίσω δεν υπάρχει οριστική συμφωνία. Το Μιστράλ είναι ένα σκάφος, ένα πλοίο το οποίο θα πουληθεί χωρίς εξοπλισμό είναι μια από τις προϋποθέσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καρδιά των συζητήσεων με τη Ρωσία και δεν διαπραγματεύεται μόνο με τη, Ρωσία, με τη Γαλλία η Ρωσία για την απόκριση αυτού του υλικού. Αντιλαμβάνομαι ότι ε, υπάρχει συναισθηματική φόρτιση σε πολλές χώρες, αλλά άλλο η συναισθηματική φόρτιση και άλλα τα συγκεκριμένα γεγονότα. Θυμήσατε κύριε Υπουργέ ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα εξαγωγή όπλων υπάρχει ένα κώδικας συμπεριφοράς που εξελίχθηκε σε κοινή θέση διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας το 2008, κώδικα συμπεριφορά ο πιο απαιτητικό στον κόσμο. Είμαστε ιδιαίτερα ενάρτητοι σε αυτόν τον τομέα και πέρα από αυτόν τον κώδικα, όπω θύμισαν συνάδελφοι, έχουμε και μια ομάδα η οποία συνεδριάζει στα πλαίσια της ΚΕΠΑ για να συζητήσει όχι μόνο την εφαρμογή αυτού του κώδικα της συμπεριφοράς αλλά και για να συζητήσει για τις εθνικές πολιτικές εξαγωγής όπλων των κρατών μελών. Υπάρχουν λοιπόν όργανα στα οποία μπορεί να συζητηθεί το θέμα των Μιστράλ με πολύ ε, ε, ουσιαστικό και συγκεκριμένο τρόπο. Αν αναφερόμαστε στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για το θέμα της εξαγωγής όπλων και στην ανάγκη να έχουμε μια κοινή στρατηγική και μια πολιτική, ε, κοινή πολιτική άμυνας πρέπει να να δούμε όλο το φάσμα του εμπορίου ε, όπλων και ε, οπλικών συστημάτων γιατί ε, ενδιαφέρει και την αμυντική βιομηχανία και νομίζω ότι πολλές χώρες πρέπει να κάνουν προόδους για να έχουμε μια Ευρώπη θέσεων εργασίας, τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και για να αυξηθεί η ικανότητά μας σε ό,τι αφορά τα στρατιωτικά μας και οπλικά μας συστήματα. Ευχαριστώ κύριε Ντοντζόν. Ο κύριος Στάλερ για 1,5 λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η εξαγωγή συγχρόνων γαλλικών ε, πλοίων στη Ρωσία έχει και πολιτική διάσταση εκτός από οικονομική. Έχει να κάνει με την αλληλεγγύη, την έλλειψη αλληλεγγύης. Αφορά τις χώρες της Βαλτικής που ανησυχούν και χώρες στην Ανατολική γειτονία τη Γεωργία, το Ζαρβαϊτζάν, την Ουκρανία και άλλες. Γνωρίζουμε ότι η Γαλλία επενεύει στο γαλλογεωργιανό πόλεμο και η Ρωσία ανέλαβε κάποιες ε, υποχρεώσεις απέναντι στη διεθνή κοινότητα. Τη στηρεί. Αφήνει άραγε τους παρατηρητές μας στη Νότια Ρωσιτία και την Απχαζία. Γνωρίζουμε ότι η κοινή θέση του Συμβουλίου του 2008 ορίζει ότι ο δικαιούχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται τις διεθνείς υποχρεώσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη. Τα κάνει όλα αυτά η Γαλλία. Η, Ρωσία, συγγνώμη, και η Γαλλία και ο πρόεδρος Σαρκοζή θα πάρει κανένα αντάλλαγμα από τη Μόσχα για αυτή την πανάκριβη αγορά. Ο κύριος Τάνοκ, για 1,5 ε, τα συμβατικά όπλα, η βιομηχανία συμβατικών όπλων αφορά πολλές χώρες και μας οδηγεί μέσα σε έναν αβέβαιο κόσμο στο να μπορούμε να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας και με αυτό μαζί με τους συμμάχους μας. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατέβαλε σοβαρές προσπάθειες για να περιορίσει την παραγωγή και την διανομή ορισμένων όπλων και να μην ε, εξάγει όπλα σε ορισμένα απολυταρχικά ε, καθεστώτα. Πιστεύω ότι οι νάρκες κατά προσωπικού είναι πολύ καλό το ότι δεν ε, χρησιμοποιούνται και αυτό αφορά και όπλα τα οποία επικρατούσαν και υπήρχαν επί ναζισμού. Αφορά και τις βόμβες διασποράς. Θα πρέπει να απομακρύνουμε τα πυρηνικά που έχουν αποθηκευτεί. Επίσης θα πρέπει να επαγρυπνούμε έναντι των τρομοκρατών που θέλουν να εισάγουν από χώρε όπου δεν υπάρχει αυστηρό καθεστώς αδειοδότηση. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει με την απαγόρευση όπλων προς την Κίνα επειδή δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και για να δείξουμε ότι υποστηρίζουμε την σύμμαχό μας, την Ταϊβάν, που βρίσκεται στην εμπροστοφυλακή ενδεχόμενης επίθεσης από την Κίνα. Βάιντερε, για 1,5 λεπτό. Κυρίες και κύριοι, τα όπλα και οι στρατιωτικά συστήματα δεν είναι προϊόν σαν οτιδήποτε άλλο. Είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια των χωρών. Η εξαγωγή όπλων σε τρίτες χώρες, κυρίως σε χώρες των οποίων το δημοκρατικό καθεστώς είναι αμφίβολο, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνεργάζονται με χώρες που υποθάλπουν την τρομοκρατία, αποτελεί μια απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες περιοχές. Γι' αυτό το λόγο αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά την εσωτερική πολιτική αλλά την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Πώς μπορούμε να μιλάμε για την ΚΕΠΑ όπως έλεγε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη στιγμή που οι χώρες μέλη πουλάνε όπλα η κάθε μία χωριστά η γαλλική απόφαση να πουληθούν πλοία Μιστράλ στην ε, Ρωσία που δεν ανήκει, μια χώρα που δεν ανήκει στην ε, στρατιωτική συμμαχία όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρωσία δεν θα πλησιάσει περισσότερο την Ευρώπη όπως έλεγε ο Γάλλος υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Καμία ευρωπαϊκή στρατηγική δεν θα στεφθεί από επιτυχία εάν παραβιάζονται ορισμένες αρχές είναι και το θέμα της αλληλεγγύης κατά την λήψη κοινών αποφάσεων. Αλληλεγγύη που υπογραμμίζεται στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρεται στον έλεγχο των εξαγωγών όπλων. Τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα δεν πρέπει να επικρατούν σε σχέση με τους αντικειμενικούς σκοπούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση που αφορά τα θέματα της ΚΕΠΑ πρέπει να εξεταστεί με όλα τα κράτη-μέλη σε συνεργασία πρέπει να εξασφαλιστεί ένας μηχανισμός νομικά δεσμευτικός και να αναλυθούν προσεκτικά όλες οι επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Όλα, αλλά, Η κυρία Γιαννάκου έχει λόγο. Για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτηση αυτή που έχει τεθεί σήμερα προς το Συμβούλιο αποτελεί ευκαιρία για να τεθεί επιτάπητος ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο είχε υποστηριχθεί από πολλούς από εμά κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής συνέλευσης αλλά και στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διάσκεψης δηλαδή η άμυνα και ασφάλεια συνολικά της ευρώπης η δημιουργία ενός οργανισμού παραγωγής όπλων και ενός κοινού αμυντικού οργανισμού. ας σημειώσουμε ότι στις ΗΠΑ παράγεται από μία γραμμή μόνο παράγονται άρματα μάχη ενώ στην ευρώπη παράγονται από 16 διαφορετικέ γραμμέ. Επομένω θα είχαμε και οικονομία κλίμακο. ωστόσο λαμβάνοντα υπόψη την κοινή θέση του συμβουλίου του 2008 για τον έλεγχο τη εξαγωγή όπλων πρέπει να ομολογήσουμε κύριε πρόεδρε του συμβουλίου ότι πραγματικό έλεγχο δεν υπάρχει. και δεν αναφέρομαι στη γαλλία αναφέρομαι σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη όπως επίσης πραγματικός έλεγχος δεν υπάρχει για το αν οι χώρες στις οποίες εξάγουμε εξάγουν σε άλλες τρίτες χώρες δηλαδή είναι ενδιάμεση, στις οποίες δεν θα θέλαμε ποτέ να δώσουμε όπλα. έχω την αίσθηση ότι η ομάδα η οποία υπάρχει στο πλαίσιο της κεπα δεν είναι σε θέση να ελέγξει τα κράτη μέλη για το πού ακριβώς εξάγουν όπλα. αν καταφέρουμε να εφαρμόσουμε την κοινή αυτή θέση και να υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί τότε θα έχουμε κάνει ένα βήμα επιτυχίας. όμως πραγματική επιτυχία στον έλεγχο της εξαγωγής όπλων θα έχουμε μόνο αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια ένα πραγματικά κοινό οργανισμό άμυνας και παραγωγής οπλικών συστημάτων που θα μας επιτρέπει να μειώσουμε το κόστος και ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε τις αρχές και τις αξίες μας δείχνοντάς το έμπρακτα στην υπόθεση και της παραγωγής και της εξαγωγής όπλων. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Δίνουμε το λόγο στην κυρία Σβένσον για 1,5 λεπτό. Και στον κύριο, με συγχωρείτε. Χτες, ο πρόεδρος της Κομισιόν στον εναρκτήριο λόγο του μίλησε για μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Μίλησε ο κύριος Μπαρόζο και για μια κοινοτική κοινή πολιτική άμυνας. Εάν δεν λάβουμε υπόψη και τον τομέα της άμυνας γενικότερα με τις εξαγωγές, τότε δεν θα επιτύχουμε τίποτα. Η συνθήκη μιλά για αρχές αλληλεγγύης και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνονται από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν πρόκειται για θέματα πολιτικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής στην ε, κοινή θέση της 8 η Δεκεμβρίου 2008 ορίστηκαν κοινοί κανόνες και τι έχουμε κάνει έκτοτε. Δυστυχώς δεν υπήρξε απήχηση αυτής της απόφασης ε, μέχρι τη Γαλλία, στη Λιθουανία και γενικότερα στις ε, βαλτικές χώρες, καθώς και στη Γεωργία. Ε, ο ναύαρχος Βλαντιμίρ Βιζότσκι είπε ότι αν οι Ρώσοι είχαν ένα μιστράλ τη στιγμή σύραξης με τη Γεωργία σε 40 λεπτά θα είχαν διευθετήσει το θέμα και όχι σε 26 ώρες. Δεν μπορεί τα μεγάλα να έχουν τέτοιες ελευθερίες. Ξέρουμε ότι θέλουν να κρατήσουν το μονοπόλιο της εξαγωγής όπλων, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Νομίζω λοιπόν ότι το Βέλγιο που έχει την Προεδρία θα πρέπει να αρχίσει τις διαβουλεύσεις για να, βρούμε, να φτάσουμε σε κοινέ διατάξεις για την εξαγωγή όπλων. Κέλαμ για ένα μισή λεπτό. you, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή έχει να κάνει με το εξή. Ε, διμερεί σχέσει των κρατών μεταξύ του απέναντι στην κοινοτική αλληλεγγύη πολίτες στα κράτη-μέλη αντισυχούν βαθύτατα για τις εξαγωγές ευρωπαϊκών κρατών στρατιωτικής τεχνολογίας σε τρίτες χώρες. Έκανε στρατιωτικές ασκήσεις η Ρωσία πέρσι στη Βόρεια Ανατολική Ευρώπη και τα σενάρια ήταν εισβολή στις βαλτικές χώρες. Και ακούσαμε τι είπε ο αρχηγός του ρωσικού στόλου ότι αν είχαμε μιστράλ ελικοπτεροφόρα στη διάθεσή μας τον Αύγουστο του 2008 θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε μέσα σε τρεις ώρες αυτή την επιχείρηση και δεν θα χάνουμε τρεις μέρες. Χαίρομαι για αυτά που είπε ο Υφυπουργό κύριος Σαστέλ. Είναι πολύ θετική ε, η αντίδραση στα μελήματα και τις ανησυχίες μας. Και ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Τανζάν που είπε ότι δεν θα πουληθεί στρατιωτική τεχνολογία. Πάντως οι Ρώσοι επέμειναν και θα συνεχίσουν να επιμένουν να αγοράσουν ακριβώς και στρατιωτική τεχνολογία. Και παραμένει προς απάντηση το εξής ερώτημα. Γιατί δεν κάνουμε διαβουλεύσεις και κανονικές συζητήσεις στο Συμβούλιο όταν θέλει μια χώρα μέλος να πουλήσει στρατιωτική τεχνολογία σε μια τρίτη χώρα. Γιατί δεν το συζητάμε αυτό και αυτό είναι μήνυμα προς το Συμβούλιο και επισήμω την προσοχή σας ότι θα πρέπει να το συζητάτε αυτό και να είναι θέμα ρουτίνας η συζήτηση αυτή στο Συμβούλιο των Εξαγωγών Όπλων Ευρωπαϊκών Κρατών προς τίτλους χώρες. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Λίζεκ για 1,5 λεπτό. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κατασκευή και εξαγωγή όπλων και στρατιωτικής τεχνολογίας είναι κάτι το οποίο είναι ένα διαχρονικό ιστορικό φαινόμενο και πάντα ε, αποτελούσε θέμα επίμαχων συζητήσεων, πάντα οδηγεί σε διχογνωμίες Υπάρχουν αλληλοκατηγορίες σε σχέση με την αποσταθεροποίηση ορισμένων περιοχών του κόσμου και ούτω καθεξής. Επίσης, ο έλεγχος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Από την άλλη πλευρά, η βιομηχανία άμυνας είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός τομέας για ορισμένα κράτη-μέλη, όπως για την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Και αυτό ισχύει και για άλλες χώρες όπως ε, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Άρα η κατασκευή και η εξαγωγή δεν θα μπορέσει στο εγγύς μέλλον να αποτελέσει αντικείμενο κοινής πολιτικής. Τα κράτη διαθέτουν μεγάλο περιθώριο ελιγμών αλλά θα πρέπει να αρκεστούν στην ε, κοινή προσέγγιση της ανακοίνωσης του Δεκεμβρίου του 2008. Η Πολωνία είχε εκφράσει πολλές ανησυχίες, καθώς και τα βαλτικά κράτη. Οι ε, ναύαρχοι της Ρωσίας ανέφεραν ότι αυτά τα πλοία μπορεί να σταθμεύσουν στην Βαλτική θάλασσα. Τώρα αρχίζει η διαδικασία Catch the Eye και δίνουμε το λόγο Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το θέμα και η προφορική ερώτηση είναι πολύ χρήσιμη. Είναι κάτι που μας απασχολεί συχνά στην Επιτροπή Εξωτερικών. Και δεν δόθηκε η ικανοποιητική απάντηση στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών. Γι' αυτό θα πρέπει το Συμβούλιο να μας δώσει μια απάντηση ουσιαστική και ικανοποιητική. Ο κύριος Κέλαμ, ο κύριος Τσαρνέσκι ε, θέτουν το ερώτημα ξανά και ξανά. Το Συμβούλιο τα συζητάει αυτά τα θέματα. Πώς γίνεται ε, αυτή η συναλλαγή δεν είναι μια απλή εμπορική συναλλαγή. Ε, είναι βαριές οι συνέπειες από την αγοραπολισία. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια οδηγία, μάλλον μια απόφαση του 2008 που ισχύει. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν ε, είμαστε προβληματισμένοι και έδειξε η υπόθεση της Γεωργίας ότι χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου. Παρακαλώ να περιορίζεστε στο ένα λεπτό. Ο κύριος Μαυρονικόλας, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομεί σήμερα μια κοινή εξωτερική πολιτική, μια πολιτική άμυνας και είναι αναμφίβολα δεδομένο ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποια πρωτόκολλα για τη συμπεριφορά στρατιωτικών βιομηχανιών απέναντι σε τρίτα κράτη. μέσα από το θέμα αυτής της συζήτησης προβάλλει όμως το δικό μου ερώτημα το οποίο νιώθω την ανάγκη να το υποβάλω στη σημερινή ολομέλεια πώς δικαιολογείται στρατιωτικές ε, βιομηχανίες και ιδιαίτερα του ηνωμένου βασιλείου να διατηρούν εμπάρκο απέναντι στην κυπριακή δημοκρατία και στις στρατιωτικές δυνάμεις της κύπρου ενώ η κύπρος είναι μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης και παράλληλα η τουρκία να δικαιούται να εξυγχρονίζει να διακινεί και να μεταφέρει εξοπλισμό και στρατιωτικό υλικό εντός των εδαφών της κατεχόμενης κυπριακής δημοκρατίας. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαυρολικόλα. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ρωμέβα. Ευχαριστώ πολύ. Είχα την ευκαιρία να είμαι συγητής του Κοινοβουλίου πριν από πολλά χρόνια και σχεδόν ομόφωνα απαιτήσαμε ο κώδικας συμπεριφοράς του 1998 να γίνει κοινή θέση, δεσμευτική, το έτος 2008. Και τότε είπαμε ότι αυτό θα είναι ένα βήμα ακόμα, αλλά όχι οριστικό. Ήταν ικανή και αναγκαία συνθήκη, αλλά όχι ικανή. Και θυμίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα Ενωμένα Έθνη υποστηρίζουν τη Διεθνή Συνθήκη για τον έλεγχο στις εξαγωγές όπλων. Αυτή είναι η ουσία. Οι εξαγωγές όπλων δεν είναι ε, σαν να εξάγει κανείς ψυγεία, ξέρω εγώ. Είναι πολύ σημαντικές οι συνέπειες γιατί τα όπλα σκοτώνουν, καταστρέφουν και ε, πτωχαίνουν κοινωνίες ολόκληρες. Όταν εξάγουμε ε, το Αφγανιστάν, στο Ισραήλ όπλα δεν είναι αθώο ε, ε αυτό. Και θα πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν είναι απλώς εσωτερική αγορά ή εμπόριο το όπλο, ή θέμα ασφαλείας και μόνο, αλλά διεθνούς ευθύνη. Και φοβάμαι ότι δεν το κοιτάζουμε από αυτή την υπεύθυνη σκοπιά. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Αντρίκινε. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε ε, βελτιώσει την συνεργασία και την αλληλεγγύη σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα την άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και την εξωτερική πολιτική. Και αυτό αφορά ιδιαίτερα την ε, περίπτωση ε, επίθεσης, επίθεση επίθεση προς ένα κράτος. Γι' αυτό η πώληση των αεροπλανοφόρων Μιστράλ φύγει ιδιαίτερα από πλευράς ε, Γαλλίας μέσα στα πλαίσια των διμερών με τη Ρωσία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με την αλληλεγγύη που προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν θα πρέπει να μειώσουμε την ασφάλεια των γειτόνων μας των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτρέπω το Συμβούλιο να κάνει ό,τι μπορεί για να συνεχίσει τη συζητήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε μια ενημερωμένη προσέγγιση πώληση όπλων σε τρίτες χώρες. Ευχαριστούμε την κυρία Αντρίκενε. Ο κύριος Τζέμπκε έχει το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα επίση την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι εξαγωγέ όπλων συνδέονται πάντα με την ε, πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξαγωγές όπλων δεν είναι ένας ξεχωριστός τομέας, ένας απομονωμένος τομέας. Κάθε συναλλαγή δεν ε, είναι απλά οικονομική ή στρατιωτική συναλλαγή, αλλά συνδέεται πάντα με θέματα πολιτικής. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να υποστηρίξω θερμά όλους εκείνους οι οποίοι ζητούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ασχοληθεί με το θέμα της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της εξαγωγής όπλων και της θετιωτικής συνεργασίας. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε πολλές αμφιβολίες σήμερα σε ό,τι αφορά την πώληση των πλοίων Μιστράλ στην Ρωσία. Αλλά αν δούμε πιο προσεκτικά αυτή την περίπτωση και αν εξετάσουμε τη δυνατότητα κατασκευής μιας αντιοπλικής ασπίδας στην Ευρώπη, θα ήταν προς το συμφέρον μας να συμμετάσχει αυτή τη διαδικασία και η Ρωσία. Πριν δώσω το λόγο στο Συμβούλιο, στον Προεδρεύοντα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Καταρίνα Νεβενταλόβα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι ειδική σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας και όπλων. Εγώ είμαι ειρηνίστρια. Θέλω να ε, εξετάσω το πρόβλημα από τη σκοπιά του Ευρωπαίου πολίτη. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατασκευάζουν οπλικά συστήματα Ε, στον κόσμο όμως υπάρχουν διάφορες σειράξεις και πόλεμοι. Και τα όπλα έχουν σχεδιαστεί για να σκοτώνουν ανθρώπους. Δεν είναι ένα προεμπόρευμα. Θα πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε από την αμυντική βιομηχανία και να προχωρήσουμε στην ειρηνευτική, αν θέλετε, ε, προσπάθεια. Και κανένας δεν μου απαντάει στις ερωτήσεις μου ε, μειώνουν την παραγωγή όπλων τα κράτη-μέλη, άραγε μήπως την αυξάνουν. Ανθεί η αμυντική μας βιομηχανία, γιατί έχουμε και οικονομική κρίση, έχουμε και υπεριστολές ή όχι. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, παρακαλώ, έχει το λόγο, ο κύριο Ελβίες Αστέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα ήθελα να επανέλθω στο τέλος της συζήτησης σε δύο έννοιες και να δώσω κάποιες διευκρινήσεις. Θα ήθελα πρώτα να επανεστιάσω το θέμα της ευθύνης. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 της κοινή θέσης προβλέπει ότι η απόφαση να γίνει ή να ε, αρνηθεί η μεταφορά ε, στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού ε, ανήκει στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. Ευθύνη ξεκινά από το εθνικό επίπεδο και η κοινή θέση βεβαίως δεν αφαιρεί αυτή την ευθύνη στα κράτη-μέλη αλλά προβλέπει μια σειρά διατάξεων που θα εξασφαλίσουν τον συντονισμό και αποτελεσματική ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών μεταξύ του. Η άλλη έννοια είναι η έννοια τη διαφάνεια, στην οποία θέλω να επανέλθω. Η κοινή θέση προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει κάθε χρόνο να ετοιμάζουν μια έκθεση για τις εξαγωγές οπλισμών τους. Μια έκθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης που ετοιμάζεται με βάση τις εθνικές εκθέσεις, δημοσιεύεται κατόπιν ετησίως και αυτή η έκθεση παρέχει στοιχεία για την οικονομική αξία των αδειών που δόθησαν με ανάλυση για κάθε κατηγορία οπλισμών καθώς και στον αριθμό των αδειών που δεν έγιναν δεκτές και αναφέρεται επίσης και στις διαβουλεύσεις που έγιναν των υστέρων μεταξύ κρατών μελών. Επίσης η ετήσια έκθεση Ευρωπαϊκής Ένωση. Εκτός από την ετήσια έκθεση, η κοινή θέση προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα δημοσιεύουν εθνικές εκθέσεις για τις εξαγωγές στατιωτικών ε, μέσων και τεχνολογία. Η, αρχή της διαφάνειας που προβλέπεται στην κοινή θέση καλύπτει σε εθνικό επίπεδο ε, ε, τα κράτη-μέλη αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολό η οποία πρέπει να δίνει και το καλό παράδειγμα. Η κοινή θέση αποτελεί όπως ορισμένοι από εσά το υπογράμμισαν άλλωστε, Μία σημαντική πρόοδο σε σχέση με τον κώδικα συμπεριφοράς. Εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2008, λιγότερο δηλαδή πριν από λιγότερα από δύο χρόνια. Βεβαίω πρέπει να αφήσουμε χρόνο στην κοινή θέση να ε, δώσει δείγματα γραφής προτού αποφασίσουμε να αλλάξουμε ε, το σύστημα και αν κατάλαβα καλά αυτά που μας είπατε, για να γίνει πιο δεσμευτικό ή να συνδεθεί με ένα σύστημα κυρώσεων. Κάτι που μπορεί να φαίνεται εγωιτευτικό. Τελευταία διευκρίνηση σε μια, σε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Η κοινή θέση, σας καθησυχάζω, συζητήθηκε κατ' επανάληψη σε πολιτικό επίπεδο, ειδικότερα στο Συμβούλιο, κυρίως στο πλαίσιο του εμπάργου κατά της εξαγωγής όπλων ή της αγοράς όπλων από την Κίνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους. Η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί στο θέμα αυτό. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι... Ναι, έχετε το λόγο. Ζητήσατε το λόγο. Ρίσ. Δεν έχω το άρθρο του κανονισμού μπροστά μου, θα ήθελα όμως να σας πω κάτι ζωτική